Good evening, dear colleagues. Uh, uh, welcome to this joint uh, Badge. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη συνεδρίαση, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, εάν συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου. Δεν έχουμε ανακοινώσει να κάνουμε, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 3, το οποίο ξέρετε πως έχει να κάνει... Um, um, ε, με μια ανταλλαγή ε, απόψεων για το θέμα ε, αυτό για το οποίο κάνουμε την κοινή συνεδρίαση με την συνάδελφο Γκαρδία Σάπαλ Ρουμπιάλ και με την Καρολίν Νακτεγκάλ. Οπότε θα ήθελα απευθεία να δώσω το λόγο σε καθέναν από τους εισηγητές και τις εισηγήτριες. Έχετε πέντε λεπτά η καθεμία για να μας παρουσιάσετε το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτά τα πέντε λεπτά να εξηγήσω ακριβώς τι έχουμε κάνει ε, με την συνεισηγήτρια και να εξηγήσουμε γιατί κάνουμε αυτή την ε, μεικτή ε, συνάντηση και γιατί δεν έχουμε σχέδιο γνωμοδότησης ή σχέδιο έκθεσης ακόμα ε, από τότε που μας διορίσατε εσείς οι ε, συγγήτριες. Παρόλο που έχουμε κάθε θέληση και κάθε βούληση να προσπαθήσουμε να βρούμε σημεία συμφωνίας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και να συντάξουμε μαζί αυτό τον κανονισμό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετά διαφορές, διαφορετικά θέσεις ε, σε σχέση με αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι ε, εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες και πάρα πολλά προβλήματα με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προσπαθήσω να ε, αποσαφηνίσω κάποια από αυτά τα θέματα και να σας εξηγήσω τι συζητάμε με τη συνεισηγήτρια και με τους υπόλοιπους συνεισηγητές. Να σας πω καταρχήν που βρισκόμαστε σήμερα. Μιλάμε για ένα κανονισμό που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, εξορισμού θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα εργαλείο για να ε, αναπτυχθούν και να εξελιχθούν οι διαστροτικές ε, αλλαγές μέσω στήριξη από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλά ερωτηματικό. Τι σημαίνει διαστροτική μεταρρύθμιση. Δεν ορίζεται αυτό κάπου και θα μπορούσαμε να περάσουμε μια ολόκληρη θητεία για το τι είναι διαρθωτική αλλαγή. Επίση, τι επιδιώκουμε μέσω αυτή τη μεταρρύθμιση. Δεύτερον, 25 δι 7 χρόνια για όλα τα κράτη-μέλη με χρήματα τα οποία θα αποδοθούν στο τέλος του προγράμματος μεταρρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Όντως, έτσι θα γίνει. Επίσης, ο πληθυσμός είναι το κατάλληλο κριτήριο για την κατανομή αυτών των ε, ποσών. Αυτό συζητάμε με τη συγγετρία αλλά οι απαντήσει που δίνουμε σε αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ διαφορετικέ. Για παράδειγμα, διορθωτική μεταρρύθμιση. Πιστεύουμε πω θα πρέπει να εντοπίσουμε το στόχο που επιδιώκουμε και να δούμε ποια είναι τα διδάγματα της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασχολείται μόνο με μακροοικονομική πολιτική και να μην κοιτάει το περιβάλλον και τα κοινωνικά θέματα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε διδαχθεί και νομίζω θα πρέπει να μπουν στο πακέτο μεταρρυθμίσεων και θα ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως 28 κράτη-μέλη. Το έχουμε πει και το λένε πάντα στους σοσιαλιστές. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να αναμορφωθεί, όπως επίσης και η ανακράτος μέλος συστάσεις. Να μπει και το περιβάλλον, γιατί χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Όχι όμως σε μόνο μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να ξεπεράσουμε τα όσα λέμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να δούμε τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη μέσα σε όλα αυτά. Δεύτερη απόκριση. Χρηματοδότηση. 25 δις είναι λίγο. Αλλά δεν έχουμε κοιτάξει το ύψο του ποσού, γιατί ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στι διαπραγματεύσει για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να αμφισβητήσουμε το ύψο του ποσού, αλλά μπορούμε να αμφισβητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή μέσω των μεταρρυθμίσεων. Γιατί ένα, σε ένα συνηθισμένο πρόγραμμα έχει προχρηματοδότηση, ενδιάμεση χρηματοδότηση και ε, τελική αποπληρωμή. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και τέλος, κλίδα κατανομή. Ο πληθυσμό ε, δεν είναι κατά τη γνώμη μου το σωστό κριτήριο. Α δούμε τι οικονομικέ περιστάσει να δούμε σε ποια θέση βρίσκονται τα κράτη αυτά, τι μεταρρυθμίσεις έχουν αναλάβει να κάνουν, ποιο είναι το εύρο των μεταρρυθμίσεων που έχουν καταθέσει για να ζητήσουν χρηματοδότηση στα πλαίσια του προγράμματο. ανεργία, παιδεία, είναι πάρα πολλά τα κριτήρια τα οποία θα ήταν ε, πιο πολύτιμα και πιο ισχυρά και όχι μόνο το πληθυσμιακό. Αυτό το οποίο λοιπόν συζητάμε αυτούς τους δύο μήνες που η Καρολίν και εγώ συζητάμε το θέμα, ε, δεν κατάφερε να μας φέρει στη χρυσή τομή. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αρχίσει και προσεγγίζουμε τις θέσεις μας και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε, ένα, σε μια έκθεση που θα βασίζεται σε έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή για να κοιτάξουμε το κείμενο. Αλλά θα επαναλάβουμε πως θέλουμε αυτή την ανταλλαγή απόψε να τη διατηρήσουμε μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Γιατί, Γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό να ξέρουμε τη θέση των υπολείπων ομάδων για τον κανονισμό αυτό. Γιατί αυτό εμπλουτίζει τη συζήτηση τη δική μας και βλέπουμε πώς εμείς όλοι μαζί στο Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσουμε μου και πέντε, το θέμα αυτό. Μου μείνα και πέντε δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην συνεισηγήτρια. Έχετε το λόγο λοιπόν συνάδελφε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Νομίζω ότι το βασικό θέμα σήμερα είναι ότι όπως προτάθηκε από την Κομισιόν στηρίζω αυτό το πρόγραμμα και δεν θα είναι έκπληξη για σας ότι υποστηρίζω και τους στόχους του προγράμματος. Τα κράτη-μέλη υλοποιούν ε, ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και αυτό θα καταστήσει ισχυρότερη την ένωσή μας και θα, αυτό θα υπερνικήσει την οικονομική κρίση. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση. Βεβαίως έχουμε συνεργασία, καλή την πίστη Υπάρχει όμως ένα χάσμα ιδεολογικό ακόμη και θα είχα προχωρήσει περισσότερο από την πρόταση της Κομισιό. Το θέμα ε, της ερεσιμότητας το θέμα της ένταξης ε, του ε, εξαμήνου ως πρόσθετο όρο. Ωστόσο, ε, ε, σημειώνω ότι αυτό πάει πέραν της πρότασης της Κομισιόν, δεν είναι κάτι το εφικτό ίσως να μπορέσουμε να έχουμε ένα τέτοιο συμβιβασμό. Έχω πέντε στόχους βασικούς, τους οποίους θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να προστατεύσω ε, το πεδίο εφαρμογής ε, της πρότασης της Κομισιόν με τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα, ευρωπαϊκό εξάμεινο, πολιτική. Είναι πρόκληση για τις χώρες να εργαστούν πάνω στα θέματα αυτά. Η συμμετοχή είναι θελοντική και τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν τις προκλήσεις ε, και το θέμα του εξαμήνου νομίζω ανταποκρίνεται στην ανάγκη των οικονομικών, των χρηματικών συνεισφορών. Και θα ήθελα επίσης να επιμείνω ότι πάνω σε αυτή τη βάση υποστηρίζω την πρώτη Κομισιόν. Δεύτερος στόχος είναι να έχουμε μια διαδικασία προσδιορισμού των μεταρρυθμίσεων που είναι επιλέξιμες για χρηματική υποστήριξη. Το πλαίσιο της Κομισιόν ρίχνει όλη την ευθύνη στην Επιτροπή. Έχουμε τις προβλέψεις, στις οικονομικές εκθέσεις, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όλη την προπαρασκευή των συστάσεων αναχώρα, ε, το πλαίσιο της πρότασης, της δεσμεύσεις μεταρρυθμίσεων και να δούμε εάν ε, θα πρέπει να γίνει μία εκταμίευση. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία χρειάζεται ε, περισσότερους ελέγχους και εξισορροπήσεις και μια συμφωνία εργαζόμαστε για την συμμετοχή περισσότερων ανεξάρτητων ε, φορέων και αυτό για κάθε χώρα μέλος. Θα πρέπει να μπορούν να εκφράσουν γνώμη για τις προτάσεις, για τις δεσμεύσεις μεταρρυθμίσεων, να είναι ένα ανεξάρτητο σώμα στην προετοιμασία των προτάσεων και να βοηθηθεί στην αξιολόγηση με τον τρόπο αυτό η Κομισιόν. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι καμιά οικονομική συνεισφορά δεν δίδεται σε κράτος μέλος που βρίσκεται στο πλαίσιο του άρθρου 7 θα πρέπει οι οικονομικές παροχές να περιορίζονται σε χώρες που τηρούν τις αξίες της Ένωσης και ξέρω ότι η τήρηση του κράτους δικαίου είναι κάτι το σημαντικό για όλους σας και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υλοποιηθεί αυτό τέταρτος στόχος θα πρέπει να δούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν προστιθέμενη αξία και ότι έχει γίνει μελέτη κόστους ωφέλους. Θα πρέπει να δίδεται χρηματοδοτική συνεισφορά μόνο για τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας και της Ένωσης. Όχι σε άλλα κράτη-μέλη. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια αξιολόγησης και νομίζω ότι από αυτό το, σε αυτό το σημείο δεν είναι ικανοποιητική πρόταση. Και πέμπτο, να διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού σύγκλησης. Θα πρέπει να έχουμε μεταρρυθμίσεις ε, που ε, ικανοποιούν τα τέσσερα κριτήρια ε, της συνθήκης ε, και επίσης ε, τηρούν την νομοθεσία της Ευρωζώνης. Βεβαίως η Οδηγία Τραπεζικής Ένωσης είναι νομίζω ένα παράδειγμα που διευκολύνει τη σύγκληση και την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν αυτές τις απόψεις για την πρόταση. Μπορούμε ίσως να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή μέσα σε ένα μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στους σκιώδεις συγητές. Ο κύριος Σαραβάμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκολτιέρη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ξεκινήσαμε με δεκάλεπτη καθυστέρηση και πρέπει να έχουμε φύγει ακριβώς 8 από την αίθουσα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε ένα μακρύ κατάλογο σκιωδών εισηγητών, ε, θα έλεγα να ε, τους ακούσουμε όλους ε, και θα ήθελα πρώτο να δώσω το λόγο στον κύριο Λαμασούρ, ε, ο οποίος είναι εισηγητής του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις τους, τις προφορικές, τις δύο εισηγήτριες. Νομίζω ότι η συντονίστρια έκον της σοσιαλιστικής ομάδας είναι εδώ. Νομίζω ότι ορισμένες ομάδες ήδη ζήτησαν ένα, ένα χρονοδιάγραμμα, διότι έχει σημασία αυτή η πρόταση και το θέμα και η αξία της ε, συνεισφοράς των εισηγητών που πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς. Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι το σύστημα που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιές, έξυπνο και οδεύει προς την κατεύθυνση μια, της ενίσχυσης της Ευρωζώνης με ικανότητες χρηματοδοτικές ή ε, οικονομικές σε σχέση με τα όσα είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν δύο σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε πρώτα απ' όλα, να αποφύγουμε το moral hazard, δηλαδή δεν θα πρέπει οι χώρες να αρχίσουν μεταρρυθμίσεις μόνο υπό τον όρο ότι θα λάβουν ενίσχυση, ότι θα λάβουν ένα ευεργέτημα. Είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα. Καλύτερα να έχουμε κίνητρα θετικά παρά κίνητρα αρνητικά. Κίνητρα αρνητικά είναι μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε για την αιρεσιμότητα, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να ανταμείβουμε μεταρρυθμίσεις που θα είναι ψευδομεταρρυθμίσεις, απλώς για να εισπραχθούν πρημοδοτήσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε μηχανισμούς γραφειοκρατικούς και βλέπουμε τις λεπτομέρειες στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα πρακτικά, τις αναφορές, τις τακτικές, ε, ενδιάμεσα στάδια, το χρονοδιάγραμμα και όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε κοινωνού, αλλά μην ε, έχουμε μια ε, γραφειοκρατία που θα είναι τρομακτική. Ευχαριστώ πολύ. για το Κυρία Μάλετιτς, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις οι διαρθρωτικές είναι πολύ επιτυχημένες ε, και πράγματι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα κράτη-μέλη γιατί προβλέπεται μια αύξηση κατά 80 εκατομμύρια ευρώ. Οφείλουμε λοιπόν να αποφασίσουμε για τη συνέχιση και την σύσταση συγκεκριμένων προγραμμάτων με στόχο να στηρίξουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη σύγκληση σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις ε, σε κεφάλαια και σε αναπτυξιακά προγράμματα. Στηρίζονται από εμά προφανώ, ε, βέβαια με διάφορα εργαλεία. Η πολιτική συνοχή είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ε, Επίση, η κοινή αγροτική πολιτική και πολλέ άλλες πολιτικές πρέπει να στηριχθούν γιατί αν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις δεν θα αποδώσουν και μακροπρόθεσμα χωρίς μεταρρυθμίσεις τελικά ε, δεν θα αναπτυχθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές απλά και μόνο ε, θα υπάρξει μία αναβολή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι ε, διαφορές και οι αδικίες ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Γι' αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για μας. Εμείς ως Επιτροπή ΕΚΟΝ οφείλουμε να στηρίξουμε το πρόγραμμα αλλά πέρα από αυτό πρέπει να αγωνιστούμε και για περισσότερες επενδύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος πυλώνας, αυτό είναι πολύ ε, καθοριστική σημασία για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Χωρίς ε, επενδύσεις ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Είναι αλήθεια ότι στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, υπάρχει μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ο συντελεστής της σύγκλησης αυξάνεται κατά 11%, 45 δις ευρώ και οι περικοπές στα ταμεία συνοχής είναι 45%. Τα νέα προγράμματα μεταρρυθμίσεων ανέρχονται σε 25 δις ευρώ ευρώ και αυτά τα 25 δις για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εκ των οποίων 2,2 δις ευρώ προβλέπονται για τη σύγκληση χωρών εκτός ευρωζώνης. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον επιμερισμό των κονδυλίων από προγράμματα μεταρρυθμίσεων ε, σε άλλα προγράμματα ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Νομίζω ότι αυτή την προσέγγιση ε, και αυτόν τον τρόπο επιμερισμού ε, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή να μην είναι καθοριστικό στοιχείο ο πληθυσμός, αλλά το περίπλοκο των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, αυτό που παίζει ρόλο είναι οι συστάσεις αναχώρα και οι μακροοικονομικές ε, ε, ανισορροπίες. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μάλατιτς ε, και λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι τόσο κακός, αλλά σας είπα δύο λεπτά για τον καθένα, κατά το μέγιστο για τους ασχελιστές. εκ μέρους της ΕΚΟΝ, του ΕΛΚΟ, ο κύριος Μαυρίτης. Θα προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ ε, σύντομος και πολύ ακριβής και να σας πω πως ε, βασιζόμαστε για αυτό το νέο πρόγραμμα ε, στο υφιστάμενο που υπάρχει για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 17-20, πρόγραμμα το οποίο μέχρι σήμερα είναι αρκετά πετυχημένο και γι' αυτό θα έπρεπε από αυτό κάπως να διδαχθούμε. Από αυτή την πρόπτικη θα καλωσορίσω την πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αλλά να σα πω πω υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτίωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτέ τι προτάσει. Καταρχήν, αν συμφωνούμε όλοι πως ο βασικός στόχος της πρότασης είναι να ε, προωθήσουμε τη σύγκληση, για να πετύχουμε ακριβώς αυτό το στόχο χρειάζεται να έχουμε κοινωνική και οικονομική σύγκληση ε, σε ισότιμη βάση. Άρα λοιπόν να προωθήσουμε και την κοινωνική σύγκληση για να προλάβουμε και να διορθώσουμε τις αρνητικές, τον αρνητικό αντίκτυπο των σφιχτών οικονομικών μεταρρυθμίσεων και να προσφέρουμε ευημερία σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, όπως επίσης και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού, που θεωρούμε πως αποτελεί ε, κομβική πρόταση που από το συγκεκριμένο πακέτο λείπει. Να σας πω λοιπόν πως από την προηγούμενη πρόταση ένα βασικό στοιχείο ήταν η ε, ενίσχυση της κατοχής του προγράμματος, κάτι το οποίο εδώ δεν το βλέπουμε και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον πρώτο πυλώνα της πρότασης, ε, τον οποίο θα πρέπει να διευρύνουμε στο πεδίο, του το πεδίο εφαρμογής και να μην περιοριστεί μόνο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τρίτον, οι μεταρρυθμίσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι φιλικές για την ανάπτυξη, με δημιουργία καλών θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να έχουμε γεωγραφική ε, σύγκληση, κοινωνική σύγκληση και ε, καταπολέμηση της ένδυας με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ένα φιλόδοξο και οικονομικά ισόρροπο και κοινωνικά ισορροπημένο πρόγραμμα έτσι ώστε μέσω της σύνδεσης με το ευρωπαϊκό εξάμεινο να τα καταφέρουμε καλύτερα. Γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν θα το πετύχουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πρέπει να τονίσω πως τα προγράμματα αυτά στήριξη μεταρρυθμίσεων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν ε, και να περικόψουν από τα όσα διαθέτουμε για την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω να είναι εδώ εκπρόσωπος της ECR για τον προπολογισμό, οπότε ο κύριος Λούκε από την ECR για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχει δυστυχώς ε, σχέδιο εκθεσής, ίσως να είναι και η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρόταση κατά περίεργο τρόπο προβλέπει πολύ ψηλό αριθμό κονδυλίων, εν πάση περιπτώσει 25 δις ευρώ, παρότι μέχρι τώρα ε, δεν υπάρχει ικανοποιητική εμπειρική ε, εμπειρία. Ε, βεβαίως υπάρχει εμπειρία με την Ελλάδα, μόνο που η Ελλάδα είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση και εφαρμόστηκε ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Τώρα, κατά πόσο αυτό μπορεί κανείς να το μεταφέρει αυτούσιο, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Απλά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια αξιολόγηση του προγράμματος. Ε, πρέπει να τεθεί το εξής ερώτημα. Βασικά, για ποιο λόγο οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να στηριζούνται από οικονομικά κίνητρα που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε τελική ανάλυση αυτές οι μεταρρυθμίσεις την ίδια τη χώρα ωφελούν. Εδώ τίθεται το θέμα της κατοχής, ένα θέμα που ακόμα δεν έχει εξεταστεί σε βάθος, όπως και αυτό που είπε και ο κύριος Λαμασούρ, το περίφημο moral hazard. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στο να υπάρξουν καθυστερήσεις ε, στις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να σας πω, εκπλήσωμαι επίσης σχετικά με τη στάθμιση των ενισχύσεων. Αυτό το Reform Delivery Tool, το περίφημο εργαλείο, θα πρέπει να ανέρχεται περίπου σε 22 δι. Βασικά, οι λογικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο, ενώ η τεχνική βοήθεια που το θεωρώ κάτι πιο σημαντικό, απλά θα προαχθούν με 48 εκατομμύρια ευρώ, μόνο 48. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή υπεραξία αυτών των προγραμμάτων. Εγώ θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή υπεραξία των προγραμμάτων προγραμμάτων θα πρέπει καταρχήν να αποδεικνύεται. Γιατί μεταρρυθμίσεις που αφορούν απλά και μόνο το ίδιο το κράτος, γιατί να πρέπει να στηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαδικασία του άρθρου 7. Καλά ακούγεται το να λέμε δεν θα υπάρχει καμία ενίσχυση, αλλά θέλω επίσης να σε επισημάνω ότι ε, κανείς δεν φταίει που καταδικάζεται αν θέλετε. Η διαδικασία του άρθρου 7 είναι σε τρεις φάσεις. Ξεκινάει μια επικοδομητική διαδικασία, διαδικασία με τη χώρα που βρίσκεται η υποκατηγορία, δηλαδή ε, με μια χώρα η οποία ακόμα δεν έχει καταδικαστεί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι στην εισαγωγή του άρθρου 7 και στις δύο πρώτες φάσεις ε, θα έπρεπε ενδεχομένω ε, να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε κύριος Μπάτ, δεν είναι εδώ αλλά εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Γκίγκολτ ε, είναι παρόν και έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους εισηγητές και θα ήθελα να πω ότι βεβαίως καταρχήν είμαστε υπέρ του Ευρωπαϊκού Εργαλείου που θα στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Αλλά για να είμαι σαφής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι θα κάνουμε εδώ, διότι μου φαίνεται ότι η περισσότερη χρηματοδότηση στο τέλος θα προέλθει από τα διαρθρωτικά ταμεία και αυτό στην πραγματικότητα στις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις ίσως ε, να προστατευτούν τα διαρθρωτικά ταμεία και στο τέλος θα έχουμε πολύ λιγότερα λεφτά από τα 25 δισεκατομμύρια που προβλέπονται για τα νέα εργαλεία, για την, την, τον ε, μηχανισμό χρηματοδότησης ε, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τη στήριξή τους. Και αυτό σημαίνει ότι στο τέλος, ίσως απλώς, ε, να έχουμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, νομίζω ότι σχετικά με τα κριτήρια υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, προβληματισμούς. Η κυρία Μαλατίτσο επίσης διαρωτήθηκε γιατί ε, να υπάρχει κατανομή κατά κεφαλή, ενώ μπορεί αργότερα τα πράγματα να είναι διαφορετικά και τα κριτήρια τα οποία έχουμε αναπτύξει με βάση την ε, συν απόφαση για τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να είναι πολύ χειρότερη για το νέο πρόγραμμα. Μπορεί ε, να μην ε, λαμβάνονται υπόψη το κλίμα, τα θέματα ισότητας φύλων με τον ίδιο τρόπο. Ας μην είμαστε αφελείς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα αποδυναμώσει τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία έχουν πολύ περισσότερες επενδύσεις και αν έχουμε κάτι ε, σαν τις νέες γραμμές θα πρέπει να έχουμε φρέσκο χρήμα. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι σχετικά με τον μηχανισμό σύγκλησης για νέα κράτη-μέλη, αυτό είναι κάτι που υποστηρίζουμε, αλλά θα θέλαμε να δούμε τα κριτήρια να είναι σαφώς ε, πέραν ε, των περιορισμών που βασίζονται στη συνθήκη, διότι το ξέπλυμα χρήματος, η έλλειψη εποπτείας, ε, υπάρχουν, αναφέρθηκε και η Τραπεζική Ένωση, όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν και οι ανισορροπίες οι μακροοικονομικές για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και στο τέλος υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με τη διαδικασία του άρθρου 7, πώς θα σχεδιάσουμε ενδολεχώς την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκίγκολτ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αφού πηγαίνουμε τόσο γρήγορα, νομίζω πως μπορούμε να επιστρέψουμε λίγο από το χρόνο σε αυτούς τους οποίους πιέσαμε τόσο πολύ, εάν θέλουν ε, να κάνουν κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις. Και κάποιοι σκιώδεις ακόμη θα μπορούσαν να μιλήσουν. Θα δώσω το λόγο τώρα. Ε, μάλλον δεν θα δώσω το λόγο στην ε, σκιώδη από την, από την ΚΟΕ. Βλέπω ότι και από την ΙΣΙΑΡ ο κύριος Διέγκο λείπει. Η FTD από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Σκιώδης, όχι. Από την Econ επίσης λείπει. Κανείς δεν είναι εδώ, οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο Catch the Eye και βλέπουμε πως έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να τα πούμε. Η κυρία Μπερές είναι η πρώτη μας ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεισηγήτριες και να σας πω πως όταν θέλει κανείς να βοηθήσει στο χαρτί τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις, συνήθως δεν ξεκινά κανεί κανείς απαγορεύοντας τον προβληματισμό και τις σκέψεις. Γιατί όταν μιλάει κανείς για διαρθρωτική μεταρρύθμιση, δυσκολευόμαστε. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε καταλάβει ποτέ και δεν έχει οριστεί ποτέ τι είναι η διαρθωτική μεταρρύθμιση. Και έχω την αίσθηση πως δεν τολμά να προχωρήσει σε ορισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μεν θα ξεκαθάριζε ε, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα στηρίξουν ή όχι τα κράτη-μέλη, αλλά θα μα έδινε τουλάχιστον ένα πλαίσιο για ε, πιο διαθρωμένου προβληματισμού, ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τι ευθύνε τη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στο τραπέζι και σήμερα μας προτείνουν ένα εργαλείο στήριξη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς περί πρόκειται. Οπότε για τη δική μου ομάδα εμείς Είπα, θα επαναλάβουμε κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ο τρόπος με τον οποίο στηρίζουμε κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά κυρίως αυτές οι οποίες στηρίζουν τα πρόσωπα, την καινοτομία, την προσαρμογή, ε, την παιδεία, ε, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Ε, αυτό θα έπρεπε να στηρίζουμε πρώτα απ' όλα αυτό που ονομάζεται κοινωνικές επενδύσεις. Και πρέπει να σας πω πως μας ανησυχεί και το πόσο θα συγκλίνουν οι οικονομίες, γιατί αυτά τα προγράμματα διορθωτικής μεταρρύθμισης απευθύνεται σε τελείως διαφορετικές οικονομίες που δεν μπορούν να συμβιώσουν ε, ε, όλες στο ίδιο πλαίσιο. Οπότε αναρωτιέμαι κατά πόσο η σύγκληση ε, συμπεριλαμβάνεται στο νέο αυτό πρόγραμμα. Έχουμε και το μικρό φάκελο, γιατί έχουμε ε, ε, το μικρό φάκελο με το μικρό ποσό για τις επενδύσεις και εκεί αναρωτιέμαι τι θα συμβεί. Δεν τολμάμε ε, να ρωτήσουμε τι θα γίνει με τα μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή και τα οποία θα στηριχθούν για να συγκλίνουμε την Ευρωζώνη. Τι θα γίνει και τι θα γίνει κυρίως μετά το Brexit. Το άρθρο 7, για παράδειγμα, πώς θα λειτουργήσει στα πλαίσια αυτού του φακέλου, τον οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε και υπό αυτό το πρίσμα για να είμαστε συνεπείς. Και πώς συνδέεται ένα τέτοιο πρόγραμμα και το γενικότερο πλαίσιο που είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τι είδους ευρωπαϊκή πολιτική στηρίζουμε, τι είδους οικονομική πολιτική στηρίζουμε. Αυτά χρειάζονται διευκρίνηση και δεν πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε οι συνεισηγήτρες εύχομαι καλή επιτυχία ε, για να καταφέρουν να δώσουν τις διευκρινήσεις που είναι απαραίτητες. Ένα λεπτό θα ζητήσω στο Catch the Eye, αλλά επειδή δεν το είπα από την αρχή, ε, σας συγχωρώ. Ο κύριος Κλίντς, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πράγματι μπορεί να είναι λογικό ε, τα διαρθρωτικά προγράμματα να συνδεθούν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Ε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε μια τεράστια γραφειοκρατία και να μην προκύψει αυτό το, αυτός ο ηθικός κινδύνος, το moral hazard. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μεταφορά κονδυλίων πρόκειται και θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα είναι προς απόλυτο όφελος τη ίδια της χώρας. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Κατά κάποιον τρόπο θα πρέπει να ισχύει το τα μέσα γιάζουν το σκοπό. Ε, καταρχήν βέβαια εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να οριστούν οι μεταρρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είτε θα γίνει με εξωτερική βοήθεια είτε με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είναι μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν σε μεγαλύτερη σύγκληση. Και οι προϋποθέσεις ε, για τις ενισχύσεις θα πρέπει να είναι πρώτον, η χώρα θα πρέπει ήδη πριν καταθέσει την αίτηση να έχει αποδείξει ότι προσπαθεί διακαώς ε, να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να επιτύχει πρόοδο. Πέρα από αυτό, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα πρέπει ε, να έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποβάθμιση από οίκους αξιολόγησης και τέλος η παράγραφος στο άρθρο υπαριθμών 7 θα πρέπει να εφαρμόζεται. Νομίζω ότι αυτό το έχουν αναφέρει και άλλοι πολλοί προλαλήσαντες. Επόμενος ε, στη διαδικασία του ΚΑΤΣΙΑ είναι ο κ. Φέμπα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά θα τον ευχαριστήσω ουσιαστικά μόνο όταν θα μας έχει καταθέσει και την έκθεση. Ε, πρέπει όμως να προχωρήσουμε λιγάκι, γιατί δεν έχει νόημα σε μία σειρά εκθέσεων ε, να έχουμε ολοκληρώσει και να καταθέτουμε και τροπολογίες, ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε καν το σχέδιο της έκθεσης. Ε, θα χαιρόμουν λοιπόν να προχωρήσουμε λιγάκι ε, με τις εργασίες μας. Δεύτερον, πραγματικά εκπλήσαμε που μιλάμε εδώ για διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Μα είναι αυτονόητο. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είναι πολύ απαραίτητε για να καταπολεμηθούν τα ελλείμματα προπολογισμών. Και διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει τι σημαίνει. Ότι μεγαλύτερα έσοδα από τι δαπάνε για να μην υπάρχει πρόβλημα όταν η χώρα θα αντιμετωπίζει ύφεση, για να έχει διαθέσιμου πόρου που θα βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί η αρνητική οικονομική συγκυρία. Αυτά είναι αυτονόητα του συμφώνου σταθερότητα. Δεν χρειάζεται χρειάζεται εδώ να συζητάμε για θέματα αρχής. Ισχύει ότι ισχύει και για την οικογένεια. Αν κανείς ζει πάνω από τις δαπάνες του, δημιουργείται πρόβλημα. Ω εκ τούτου και τα κράτη ε, οφείλουν μακροοικονομικά να κάνουν ακριβώς το ίδιο, διότι οι μεταρρυθμίσει και αυτέ είναι δαπανηρές. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε πάνω στο μηχανισμό που θα πρέπει να εφαρμόζουμε, νομίζω θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ο κύριος Γκέρολτ έχει το λόγο. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας στο άρθρο 16 παράγραφος 1 Εκεί προβλέπεται μία περίοδο ε, πέντε ετών ε, για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Εγώ αυτό το βρίσκω μικρό, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί ξέρετε κάτι, εν μεταξύ έχει αποδειχθεί ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κυβερνήσει οι οποίε ε, με το που αναλαμβάνουν τα ενία δεν προβαίνουν σε μεταρρυθμίσει Και μόνο αυτό, αλλά έρουν και μεταρρυθμίσει που είχαν δρομολογηθεί από προηγούμενε κυβερνήσει. και λένε μα εμεί δεν δεσμευόμαστε. Εξ όσων γνωρίζω, για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, εγώ θεωρώ ότι το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Παράγραφος 16.1, εκεί γίνεται λόγος για 10 χρόνια και αυτό πρέπει να πω κατά κανόνες συμπίπτει με δύο θητείες. Και έτσι καλύπτουν δύο ή και τρεις περίοδοι, κυβερνητικές περίοδοι. Είμαι πεπισμένος ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων και θα ήθελα να παρακαλέσω τους και ηγητές να λάβουν υπόψη τους αυτή τη δική μου πρόταση. Πολύ ωραία. Ο τελευταίος που ζητά το λόγο, ο κύριος Καλβέ. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικές επιπτώσεις ε, σημαντικές από το κείμενο. Ε, αυτό συμβαίνει πάντα σε τέτοιες προτάσεις. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Απασχόλησης αποφάσισε να μην καταθέσει γνωμοδότηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όσο μου συντονιστής για την Επιτροπή Απασχόλησης, παίρνω το λόγο για να μιλήσω στις ε, συνεισηγήτριες και να τους πω να, να παρακαλέσω μάλλον να κάνουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να βρουν ένα κοινό τόπο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για να δημιουργήσουμε αλληλεγγύη που θα είναι αποτελεσματική και συνοχή η οποία θα δημιουργήσει αυτή την αίσθηση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και λέω το εξής. Μου φαίνεται πως το να πούμε πως ένα κριτήριο θα είναι το πληθυσμιακό και θα ε, δώσουμε περισσότερα χρήματα σε όσους έχουν ε, μεγαλύτερο πληθυσμό είναι τουλάχιστον ανεκδότο. Ευχαριστώ και πριν δώσω το λόγο πίσω στον κύριο Γκαλτιέρη και να του δώσω και την Προεδρία, σας ρωτώ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Έχουμε ένα μικρό περιθώριο. Κανείς. Κύριε Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα αναφερθώ σε μερικά από τα σημεία ε, που αναφέρθηκαν το θέμα του πληθυσμού. Γιατί η Επιτροπή έχει ε, μιλήσει για αυτό το δικαίωμα κατανομής. Τα κίνητρα, τα οικονομικά είναι ανάλογα με το μέγεθος της χώρας για να υπάρχει ένα πραγματικό κίνητρο. Πρέπει να ε, υπάρχει μια συνεισφορά αρκετά σημαντική και πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των διαθεσίμων πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το κριτήριο λοιπόν με βάση το πληθυσμό ανταποκρίνεται στις δύο αυτές ανάγκες. Πρώτον, να υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο ε, σε όλες τα κράτη-μέλη για να γίνεται αίσια η διαδικασία και να επιτρέπεται σε κάθε ε, πολίτη να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλεονέκτημα και χρήματα από αυτό το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να επαναλάβω ότι το θέμα αυτό του ε, πληθυσμού βασίζεται στην νομική βάση για την πολιτική συνοχή. Η νομική βάση του προγράμματος είναι 105.3 που είναι το θέμα της συνοχής και υπάρχουν και άλλους, άλλοι μηχανισμοί γνωστοί σε όλους μας, ε, το Ταμείο Αλληλεγγύης και λοιπά που έχουν την ίδια νομική βάση και βασίζονται σε μια κατανομή, μια κλίδα κατανομής ουδέτερη Λοιπόν, δεν κάνουμε κάτι το οποίο είναι αντίθετο προς το θέμα της συνοχής, την ανάγκη να υπάρχουν θέματα ε, περιβαλλοντικά, κοινωνικά που να ενσωματωθούν. Αυτό είναι εφικτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι ένα πρόγραμμα εθελοντικό, βασίζεται σε πρωτοβουλία των κρατών μελών και η επιλεξιμότητα των ε, μεταρρυθμίσεων είναι, γίνεται βάση των συστάσεων αναχώρα, ε, και το περιβάλλον το μακροοικονομικό, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Κομισιό των, που σχετίζονται με τα κράτη-μέλη και αυτά τα έγγραφα τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Κομισιόν πάνε πέραν θεωρητικά από το, την απλή ε, πειθαρχία, την δημοσιονομική, τη μεταρρύθμιση σχετικά με την πειθαρχία, τα θέματα περιβάλλοντος και άλλα θέματα, τα κοινωνικά θέματα εξορισμού είναι επιλέξιμα βάση του προγράμματος. Σχετικά με το moral hazard, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχετε βεβαίως προβληματιστεί για το πώς ε, να αποφύγει κάτι που θα οδηγήσει στο moral hazard. Οι λύσεις τις οποίες προτείναμε βασίζονται στο γεγονός ότι οι αναφορές από τα κράτη-μέλη, οι εκθέσεις είναι στο ευρωπαϊκό εξάμεινο συντονισμού της οικονομικής ε, πολιτικής. Υπάρχει εξέταση από και το γεγονός ότι το πληρωμή γίνεται μόνο στο τέλος με βάση το στόχο και ούτως αυτό γίνεται ούτω ώστε να αποφύγουμε το moral hazard, γίνεται η πληρωμή στο τέλος, διότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο κίνητο, υλο, κίνητρο υλοποίηση ε, των μεταρρυθμίσεων και για να μην γίνει καμιά μεταστροφή ε, ενδιαμέσως. Ένα άλλο θέμα, η σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, βεβαίως είναι τα δύο αυτά προγράμματα, τόσο τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων είναι κάτω από το κεφάλαιο της συνοχής, είναι συνδεδεμένα και τα δύο υπάρχει μια συμπληρωματικότητα που πρέπει να αξιοποιηθεί, υπάρχει μια διαχωριστική ε, γραμμή. Ε, έχουμε την μία που σχετίζεται με τις επενδύσεις, ε, με το φυσικό κόστος, το υλικό κόστος των επενδύσεων ενώ το εργαλείο θα ασχοληθεί ε, με τις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το μηχανισμό συντονισμού που υπάρχει στο επίπεδο της Επιτροπής σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ε, ο κύριος Γκίγκολτ νομίζω θέλει να λάβει το λόγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να κάνετε μία παρατήρηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω μόνο να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως ε, θα έπρεπε να απαντήσει και σε όλα τα άλλα ερωτήματα. Δυστυχώς τα γνώρισα, αλλά όλοι οι άλλοι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν επ' αυτόν. Και πρέπει να σας πω, δεν είμαι ακόμα πεπισμένος γιατί η γερμανική κυβέρνηση να πάρει 4 δις ε, ευρώ έξτρα και υποτίθεται θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις και δεν θα είναι μόνο 4 δις. Εγώ ε, έχω υπολογίσει ότι αν τελικά δεν μείνει η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία θα πάρει πέντε δι. Γιατί να πρέπει η Γερμανία να πάρει πέντε δι ω παρολογικό κίνητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διάσταση την κοινωνική και την περιβαλλοντική στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο την έχει υποβαθμίσει, την έχει αμβλύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί και αυτή υποβαθμίζει αυτά τα κριτήρια στις συστάσεις ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί να πρέπει να δεχθούμε αυτή την όθευση, αυτή την ε, υποβάθμιση των κριτηρίων σε σχέση με την χορήγηση των κονδυλίων, ενώ ε, στα κανονικά διαρθρωτικά ταμεία διατηρούμε αυτά τα κριτήρια. Παρακαλώ, αν έχετε το λόγο να απαντήσετε, ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Γιατί η Γερμανία να πάρει όλα αυτά τα χρήματα, κοιτάξτε, η απάντηση είναι ότι ε, στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται άμεση καταβολή στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα σύστημα αρκετά καινοτόμο, θα το χαρακτήριζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σχέση με τη μέγιστη οικονομική συνεισφορά. Άρα δηλαδή αν ένα κράτος μέλος προτείνει μεταρρυθμίσεις ε, στο πλαίσιο του προγράμματος και αν υπάρχει στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης θετική αξιολόγηση και οι μεταρρυθμίσεις ε, εφαρμόζονται και υπάρχει και ο πληθυσμός. Εκεί ισχύει το 50% καταβολή ενισχύσεων και Δηλαδή κανένα κράτος μέλος δεν ε, δικαιούται εξ ε, να λάβει αυτά τα προγράμματα. Αν δεν τα πάρει ένα κράτος αυτά ε, τα χρήματα θα πάνε ε, σε ένα κοινό κορβανά που θα είναι διαθέσιμο σε, για όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, για την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση, δεν είναι ότι αποκλείονται ε, μπορούν να ενταχθούν μέσα στο πρόγραμμα, στο βαθμό βέβαια που τα κράτη-μέλη καταβάλουν σχετικές προτάσεις που έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή προφανώς με το, με το περιβάλλον. Ευχαριστώ λοιπόν. Ποιο θέλει να ξεκινήσει από τι ε, συγγήτριε, να δώσουμε το λόγο με την αντίστροφη ε, σειρά. Η συγγήτρια από τους φιλελευθέρους λοιπόν πρώτη. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σας αγαπητοί συνάδελφοι και νομίζω ότι ένα συνάδελφος είπε συμφωνούμε επί της αρχής και αυτό είναι το ο πυρήνας του θέματος. Θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι όλοι θα πατήσουμε πως ναι. Και αυτή είναι η αρχή που διέπει την πρόταση και γι' αυτό θεωρώ και από τις αντιδράσεις σας πως υπάρχει στήριξη για το πρόγραμμα, αλλά υπάρχει και η εξή ερώτηση. Με ποιο τρόπο θα γίνουν καλύτερα τα πρόγραμματα αυτά και θα ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ακούω λοιπόν για τον ηθικό κίνδυνο, το moral hazard, το είπε ο κύριος Λούκη, ο κύριος Λαμασούρ, το ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ απολύτως, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του προγράμματος. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση για το πεδίο εφαρμογή. Κατανοώ γιατί κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά η χρήση του πεδίου εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου εξασφαλίζει πως μόνο οι ουσιώδεις και συνολικές σφαιρικές μεταρρυθμίσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και γι' αυτό θέλω να διατηρήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ως στόχο. Τέλος, κατανοώ γιατί όλοι περιμένουν την έκθεση και νομίζω πως και οι συνάδελφοι και εγώ θέλουμε να κλείσουμε την έκθεση και η ανταλλαγή απόψεων μας πιέζει να κλείσουμε το θέμα, αλλά μας δίνει και περισσότερες μια καλύτερη καθοδήγηση, οπότε μέχρι τα τέλη του μήνα ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Η Aider. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο που μας ε, εξήγησαν ποιες είναι οι απόψεις τους για τον κανονισμό αυτό και που προσθέτουν στοιχεία στη συζήτηση η δυσκολία που έχουμε με την συνεισυγήτρια για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σε ελάχιστο παρανό... παρανομαστή είναι μία προσπάθεια που θα οδηγήσει στο να ακουστούν όλες οι απόψεις που εξέφρασαν οι πολιτικές ομάδες εδώ. Είμαστε πολύ εργατικές και θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να πετύχουμε μία συμφωνία έτσι ώστε να παρουσιάσουμε σε εσάς ε, αυτή την έκθεση. Δύο σχόλια. Για τον ηθικό κίνδυνο να σας πω πως με εκπλήσει το ότι όλοι μίλησαν για το moral harass. Αν δούμε την κατανομή των ε, κονδυλίων ανακρατός μέλος, δεν θεωρώ, δεν θεωρώ α, ε, πως η Γερμανία θα πάψει να κάνει μεταρρυθμίσεις για τα δύο δις. Είναι δύο δις, όχι τέσσερα, ή η Γαλλία ή η Ισπανία. Δεν νομίζω πως υπάρχει οποιοδήποτε ηθικός κίνδυνος για οποιαδήποτε χώρα ε, και ότι θα σταματήσουν τις μεταρρυθμίσεις περιμένοντας να τους στείλουμε αυτά τα χρήματα, νομίζω ότι θα μπορούσαν να έχουν και 10 φορές παραπάνω χρήματα και πάλι αυτό να μην τους ε, αποτρέψει. Αυτά, περιθικού κινδύνου. Και δεύτερον, ορισμός των ε, διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Τι είπε ο κύριος Φέρμπερ. Ναι, είναι για να ξεπεραστούν τα διαρθωτικά προβλήματα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ορισμός, αλλά αν δούμε τι λέει η ΕΚΤ, για τη διαστρωτική μεταρρύθμιση, ο ορισμός εκεί είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Η ΕΚΤ, που νομίζω πως δεν είναι ε, πολιτικά προοδευτικό όργανο, μιλά για ισορροπημένη ανάπτυξη που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η ισότητα και η πρόσβαση στην παιδεία, στην ε, υγεία που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική ευημερία. Άρα λοιπόν, ανάλογα με την οπτική γωνία που έχει ο καθένας μας, ε, δημιουργεί δυσκολίες στο να αποφασίσουμε ποια είναι τα κριτήρια και οι στόχοι στο πρόγραμμα. Αλλά μην χάνουμε το χρόνο μας προσπαθώντας να βρούμε ε, ε, ορισμούς. Ας συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα κοινό τόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας καταθέσουμε, όπως σας είπα, αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχόμαστε πολύ επιτυχία στην εργασία σας. Η προθεσμία για τις τροπολογίες θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. Είναι το τέλος του σημείου 3. Έχουμε το 4, διάφορα, 5, Έχουμε με την πέμπτη το πρωί, την 8 το πρωί με την Επιτροπή Προϋπολογισμού, όχι σε αυτήν την αίθουσα, αλλά έναν όροφο το ΒΙΚ 100, θα συζητήσουμε ε, την, ε, την EISF, τον μηχανισμό των σταθεροποιητικών. Ευχαριστώ πολύ. Λύε τη συνεδρίαση.